Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο θα βρούμε το σωστό τρόπο να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ θερμά κύριε Επίτροπε. <clears throat> Λίγη συζήτηση αυτή τη έκθεση. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση τη κυρία Γκρουνή. Άτυπε συμβάσει, εξασφαλισμένη επαγγελματική πορεία και νέε μορφέ κοινωνικού διαλόγου. Το λόγο έχει η συγγήτρια για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι. Ένα μήνυμα πρέπει να συγκρατήσουμε όλοι ότι οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης αορίστου διαρκείας πρέπει να είναι ο κανόνας και γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε απογοητευμένοι γιατί ένα τέτοιο θέμα που είναι στα πλαίσια της στρατηγικής 2020 να μην γίνει αντικείμενο συζήτησης. Πολλοί συνάδελφοι θα ήθελαν να μιλήσουν αλλά δεν είχαν την δυνατότητα. Τους ζητώ όμως να συνεισφέρουν γραπτά τις ιδέες τους. Συνεργαστήκαμε με όλες τις πολιτικές ομάδες, καταλήξαμε μετά από αρκετές διαβουλεύσεις σε μια συμφωνία και μια, ένα, ένα εναλλακτικό ψήφισμα κατετέθη από τους πρασίνους. Αυτά που προσθέτει η κυρία Σρέτερ στο εναλλακτικό της ψήφισμα δεν μπορούν να υποστηριχθούν από την δική μου ομάδα και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή της είχε έτσι και αλλιώς καταψηφίσει. Επί της ουσίας των προτάσεων αυτό για τους ψευδο ανεξάρτητους εργαζομένους. Πράγματι η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί αποκτά διαστάσεις μάστιγας. Είναι σαφές ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε καλύτερους ορισμούς για τους ανεξάρτητους εργαζομένους και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα σωστά κριτήρια. Ο ορισμός που προτείνουν οι πράσινοι είναι εντελώς θολός και δεν προσφέρει τίποτα στην κατανόηση του προβλήματος. Τώρα, σχετικά με την επίκληση μιας οδηγίας που να εγγυάται τα ίδια δικαιώματα των εργαζομένων, το δικαίωμα του να ανήκουν σε συνδικάτο ανεξαρτήτως επαγγελματικού καθεστώτος. Για ποιο δικαίωμα μιλάμε τώρα και ποιος εμποδίζει τους ανεξάρτητους εργαζομένους να συνδικαλίζονται. Νομίζω ότι η επίκληση συγκεκριμένης οδηγίας είναι εκτός κοινοτικών αρμοδιοτήτων. Στην έκθεσή μου, θέλησα να καταστήσω το συγκεκριμένο αυτό τρόπο απασχόλησης τον κανόνα και να μην αντικατασταθούν από ατυπικές μορφές απασχόλησης. Υπενθυμίζω ότι η αρχή της ελαστασφάλειας είναι κάτι το οποίο στοχεύει κυρίως στην διασφάλιση του εργαζομένου και αυτό δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να παραβιαστεί σαν αρχή δεν θα πρέπει να μειώσουμε τι επενδύσει που θα οδηγήσουν σε μόνιμες θέσει απασχόλησης. Δυστυχώ τα ποσοστά ανεργία είναι υψηλότατα και οι ατυπικές μορφές συμβάσεων δυστυχώ αυξάνονται συνεχώ. Στους νέους τα ατυπικά αυτά συμβόλαια μπορεί να είναι ίσως μια πρώτη επαφή με την αγορά εργασίας. Αν κάτι τέτοιο δώσει μια δυνατότητα στου νέου και οδηγήσει σε μια πρόσληψη με αόριστο χρόνο, γιατί και όχι αν μπορούμε να αποφύγουμε έτσι μακρές περιόδους θα έλεγα αδράνειας επαγγελματικής. Τέλος, αν αυτή η ατυπική μορφή ε, εργασιακής σχέσης είναι μεταβατική, όταν περνάει κανείς σε μια εντελώς διαφορετική μορφή απασχόλησης, γιατί όχι για μια ακόμη φορά. Σημασία έχει να κρατήσουμε τον εργαζόμενο στην αγορά εργασίας. Επιμένω επίσης στον βασικό ρόλο που παίζουν οι κοινωνικοί εταίροι και οι εκπρόσωποι της κοινωνίας της αγοράς στην επεξεργασία και την εφαρμογή των πολιτικών απασχόλησης. Απευθύνω έκκληση σε όλα τα κράτη-μέλη να εμπλέξουν τους νέους όσο και περισσότερο γιατί μέχρι τώρα ποικίλουν οι παρεμβάσεις των διαφόρων χωρών. Θα πρέπει να προχωρήσουμε στην κοινωνική συνοχή επίσης. Μέσω της εκθέσεως αυτής το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα κράτη-μέλη και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η σωστή διαδικασία ελέγχου της κοινωνικής και εργασιακής εξέλιξης είναι κάτι το απαραίτητο. Ελπίζω το Συμβούλιο να σεβαστεί τις αποφάσεις τις οποίες είχε πάρει στο παρελθόν. Έχουμε ανάγκη από ξεκάθαρου προσανατολισμούς και συγκεκριμένα μέτρα για να διατηρήσουμε τι θέσει απασχόλησης στις περιφέρειές μας και να ανοίξουμε νέες προοπτικές στα πλαίσια της στρατηγικής 2020. Τέσσερι αιτήσει για τη διαδικασία Καστιάη. Ναι, ναι, όχι, όχι, όχι, ναι, όχι. Κύριε Ρώση, σας έχω καταγράψει. Κέστιγκερ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την έκθεση αυτή γιατί έχει μια επίκαιρη μορφή προβληματισμού για την αγορά εργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ευελίξη ασφάλεια δείχνουν οι στατιστικές τα τελευταία χρόνια ότι υπάρχει μια μεγάλη μετατόπιση προς την προσωρινή εργασία στην ευρωπαϊκή αγορά. Και όχι μόνο αυτό, οι ατυπικές μορφές εργασίας έχουν αυξηθεί. Αυτό αφορά ιδίως την απομείωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Και δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή είναι σε κίνδυνο πολλές θέσεις εργασίες, υπάρχει όλο και μεγαλύτερη κατάξυση αυτών των ατυπικών μορφών εργασίας. Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό χρειάζεται μια σαφής γραμμή πλεύσης αυτή αναφέρεται και στην έκθεση της κυρίας Γκρίνη. με τη δημιουργία θέσεων εργασίας οι οποίες είναι αηφόρες, με την πρόθεση της κατάρτισης, με την εξασφάλιση ισότητας ανδρών και γυναικών. Όλα αυτά αναφέρονται στην έκθεση της κυρίας Γκρινή. Θα πρέπει λοιπόν η ευέλικτη ασφάλεια να μην χρησιμοποιηθεί για να υπονομεύσει περισσότερε θέσει εργασία. Ευχαριστώ. Κομφεράτη. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Γκρουνή, όχι μονάχα για τη θαυμάσια εργασία που έχει φέρει σε πέρας, αλλά και για τη μεγάλη ευαισθησία που έχει επιδείξει, λαμβάνουν υπόψη και την άποψη των άλλων πολιτικών σχηματισμών. Είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται πολύ συχνά και γι' αυτό θέλω να το υπογραμμίσω. Υπάρχουν ορισμένες ιδέες οι οποίες αναφέρονται στο έγγραφο της κυρίας Γκρούνη ότι θα πρέπει η εργασία περιορισμένη διάρκεια να θεωρείται σαν κανονική εργασία σε ό,τι αφορά την προστασία των εργαζομένων. Είναι απαραίτητο λοιπόν να μπορούμε να έχουμε σε ορισμένε περιπτώσει ανθρώπου με σύμβαση περιορισμένου χρόνου, αλλά θα πρέπει να έχουν ακριβώ τα ίδια δικαιώματα όπω και οι άλλοι εργαζόμενοι. Αυτό θα οδηγήσει σε μια ομαλοποίηση των σχέσεων εργασία χωρί ιδιαίτερη επισφάλεια. Αλλά επίση είναι σημαντικά αυτά τα οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη για το κοινωνικό διάλογο. Να κατανοήσουμε ποια είναι η σημασία τη εκπροσώπηση και των εργοδοτών και των εργαζομένων. Οι συλλογικέ συμβάσει και η συλλογική εκπροσώπηση είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο <clears throat> τη κουλτούρα στον εργασιακό τομέα που θα οδηγήσει και σε μεγαλύτερη συνοχή στη σχέση εργαζομένων και εργαδοτών. για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πίεση για όλο και μεγαλύτερη ευελιξασφάλεια, <clears throat> όπως λέγεται, έχει οδηγήσει στην αύξηση και στον πολλαπλασιασμό των θέσεων εργασίας, επισφαλών θέσεων εργασίας. Έτσι τροποποιείται το σύνολο σχεδόν των θέσεων εργασίας σε θέσεις οι οποίες είναι ατυπικές και καλύπτονται από αυτή την περίφημη ενέργεια της ευελίξης αυτό οδηγεί και σε μία αύξηση της απασχόλησης. Αυτό είναι χαρακτηριστικό της τωρινής όξυνσης των συνθηκών του καπιταλισμού και οδηγεί στην εξαθλίωση των εργαζομένων γιατί είναι τόσο χαμηλές οι αμοιβέ τους που δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ζήσουν με αξιοπρέπεια. 9 εκατομμύρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν το 2008 ήδη οι άνεργοι και τώρα είναι πολύ περισσότερα τα εκατομμύρια αυτών που ζουν σε συνθήκες ένδυας και εξαθλίωσης παρά το γεγονός ότι εργάζονται. Χρειάζεται λοιπόν μια ρήξη με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές οι οποίες έχουν υπονομεύσει τα εργασιακά δικαιώματα όπως και με την ιδέα της ευέλικτη ασφάλεια. Πρέπει να την αντικαταστήσουμε με την αξιοπρέπεια στην εργασία που μόνο αυτή δημιουργεί πλούτο. Κύριος Ρώση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να συνεχίσω με αυτά τα οποία έλεγε η προηγούμενη συνάδελφος. Οι χαμηλές αμοιβέ εμποδίζουν την κυκλοφορία του χρήματος. Στην ουσία αυξάνει η ένδυα και αυξάνονται και οι δυσκολίες. Αυτές οι ατυπικές μορφές απασχόλησης ναι μεν αυξάνονται, αλλά αν χρησιμοποιηθούν έξυπνα μπορεί να βοηθήσουν κοινωνικά. Για να το πετύχουμε θα πρέπει να σεβαστούμε ορισμένες προϋποθέσεις να συνδυάσουμε την ευελιξία με την ασφάλεια και να αποφύγουμε καταστάσεις όπου εργαζόμενοι χωρίς προσόντα παίρνουν συστηματικά θέσεις χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις με ελάχιστες αμοιβέ. Όλα αυτά συνδέονται με την κατάρτιση διαβίου των εργαζομένων. Μόνο αυτό θα δώσει εγγυήσεις για την κοινωνική επανένταξη των απολυθέντων εργαζομένων και μπορεί να βοηθήσει μια τέτοια μορφή ατυπική απασχόλησης και στην καταπολέμηση της φεάς εργασίας που μαστίζει τις οικονομίες μας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και πάλι ευχαριστώ την εισηγήτρια κυρία Γκρούνη για την έκθεσή της που είναι και πολύ επίκαιρη Βλέπω ότι τα οργανώσατε με τρόπο ώστε τα θέματα να συσχετίζονται μεταξύ τους. Τα θέματα που θίγει εδώ η κυρία εισηγήτρια στην έκθεσή της είναι όντως επίκαιρα διότι τα ατυπικά συμβόλαια, τα μη συνήθη συμβόλαια είναι κάτι που είναι προβληματικό και θα έπρεπε να λυθεί για να δημιουργηθούν κατάλληλες συνθήκες εργασίας στην αγορά. Ένα από τα κυριότερα μηνύματα της έκθεσης που δέχομαι γιατί συμφωνεί με τη γενικότερη γραμμή της έκθεσης ε, είναι ακριβώς ένας από τους στόχους του προγράμματος 2020. Οι αρχές της ασφαλιξίας ή ευελιξασφάλειας είναι κάτι το οποίο μπορεί να αποτελέσει ένα μοχλό αντιμετώπιση της κρίσης. Πρέπει παρά το ότι όλοι δέχονται την αρχή αυτή να αλλάξει ο τρόπος εφαρμογής της έχοντας πάρει μαθήματα από την κρίση που οδήγησε σε μεγαλύτερη ανεργία και την απέτηση για όλο και μεγαλύτερες αλλαγών στις θέσεις εργασίας του καθενός και της καθεμιάς. Η ασφαλιξία πρέπει να ενισχυθεί σε όλα τα επίπεδα απασχόλησης και σε επίπεδο ολόκληρων επιχειρήσεων. Αυτό είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση. Η Κομισιόν θα στηρίξει θα υποστηρίξει την εφαρμογή του προγράμματος Ευρώπη 2020 μέσω ορισμένων πρωτοβουλειών, μία από τις οποίες ανέφερα προηγουμένως. Μία δεύτερη θα συμπεριλαμβάνει ένα ολόκληρο πρόγραμμα εργασίας για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, για τους νέους ακριβώς, για τους νέους τα επόμενα χρόνια. Η πρόταση αυτή που θα υποβληθεί τον Νοέμβριο στοχεύει στη δημιουργία συνθήκων εξυγχρονισμού της αγοράς εργασίας, αύξησης του ρυθμού της απασχόλησης και βιωσιμότερης ανάπτυξης των κοινωνικών μας προτύπων. Θα καλύπτει πολλά από τα θέματα που θίγει και η κυρία Γκρουνίου όπως την ευελιξασφάλεια ή ασφαλιξία και τον κοινωνικό διάλογο. Κυρία Γκρούνη, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι βουλευτέ, η Κομισιόν και εγώ ο ίδιος προσβλέπουμε με μεγάλη αδημονία στις επόμενες συζητήσεις μας του θέματος αυτού. Ευχαριστώ. Ε, η ψηφοφορία θα διεξανθεί αύριο στις 12 το μεσημέρι. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση του κυρίου Φερνάντε, πράσινη βίβλο τη Επιτροπή για τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το λόγο έχει ο εισηγητή για τέσσερα λεπτά.